σύμφωνα με το άρθρο 4 της παραγράφους 1 και 3 του κανονισμού σύμφωνα με την παράγραφο 4 του κανόνα 231 ε, ψηφίζουμε το κείμενο το οποίο θα βρείτε στο σελίδα της Ολομέλειας. Σύμφωνα με το άρθρο 78 ε,